Παρακαλώ τους δημοσιογράφους να τελειώσουν τη δουλειά τους και να μπορέσουμε έτσι να αρχίσουμε. Θα σας δώσω 15 δευτερόλεπτα ακόμη και μετά θα πρέπει να αποχωρήσετε, κυρίες και κύριοι του τύπου. Παρακαλώ μην καταλάβετε θέσεις που σαφώς προορίζονται για άλλους. Υπάρχει και χώρος ακρόασης, αίθουσα ακρόασης όπου μπορείτε να παρακολουθήσετε. Υπάρχει επίσης και η μετάδοση από το διαδίκτυο. Θα παρακαλέσω, λέει ο πρόεδρος κ. Σκουαλτιέρη, θα παρακαλέσω τις και τους δημοσιογράφους να αποχωρήσουν. Μην κάθεστε παρακαλώ μπροστά από τους βουλευτές. Please. We have to start our... Πρέπει να αρχίσουμε την ακρόαση, παρακαλώ. So, good afternoon to everyone. Καλό απόγευμα σε όλου και όλου. Θα ήθελα πρώτα να απευθύνω το καλό ορίσατε στον υποψήφιο επίτροπο κύριο Χιλ για την ακρόαση ενώπιον της Επιτροπής Οικονομικών. Γνωρίζετε ότι σκοπός της ακροάσεως είναι να επιτρέψει στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ασκήσει τα δικαιώματά του που απορρέουν από την συνθήκη για την ακρόαση του Επιτρόπου και να μπορέσει η Κοινοβουλευτική Επιτροπή να αξιολογήσει εάν το προτινόμενο πρόσωπο, ο υποψήφιος Επίτροπος, είναι κατάλληλος να γίνει Επίτροπος αλλά και να ασκήσει και τα καθήκοντα που απορρέουν από το χαρτοφυλάκιο του. Σύμφωνα με τους σύμφωνα με τον κανονισμό του Κοινοβουλίου, άρθρο 16, το Κοινοβούλιο αξιολογεί τον υποψήφιο επίτροπο στην βάση των γενικών του ικανοτήτων, ε, της ευρωπαϊκής του δέσμευσης, των γνώσεων, ε, των θεμάτων του χαρτοφυλακίου του, των επικοινωνιακών του δεξιοτήτων, πολιτικών προτεραιοτήτων και της γενικής συμβολής του στο έργο της νέας Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Υπενθυμίζω επίσης ότι πριν την ακρόαση ο υποψήφιος επίτροπος έχει απαντήσει ήδη γραπτός σε ερωτήσεις του προπαρασκευαστικού ερωτηματολογίου και οι γραπτές απαντήσεις του έχουν διαβιβαστεί σε όλες τις γλώσσες στους ευρωβουλευτές. Σύμφωνα με την προβλεπόμενη διαδικασία έχει καταθέσει και δήλωση περί των συμφερόντων του και η αρμόδια κοινοβουλευτική επιτροπή δεν έχει καμία ένσταση. Τώρα, επιτρέψτε μου να εξηγήσω την ε, δομή της συζητήσεως. Θα προσκληθεί πρώτα ο υποψήφιος επίτροπος να προβεί σε, γραπτή, σε, συγγνώμη, σε προφορική δήλωση έως 15 λεπτών και διαθέτει και 5 λεπτά στο τέλος ε, της ε, ακροάσεως για μια καταληκτική δήλωση. Μετά από την πρώτη εισαγωγή έχουμε 45 ερωτήσεις με σλότ τριών λεπτών, ε, ένα λεπτό υποβολή ερωτήσεως ή δύο λεπτά απάντηση. Πρώτα θα ε, ερωτήσουν οι εκπρόσωποι των πολιτικών ομάδων και οι μη εγγεγραμμένοι για να μπορέσουν να θέσουν τις ερωτήσεις τους όλοι οι βουλευτές θα επιμείνω αυστηρά στην τήρηση του χρόνου των τριών λεπτών και θα είμαι υποχρεωμένο να αφαιρέσω τον λόγο από τον Ευρωβουλευτή που ενδέχεται να ξεπεράσει τον χρόνο του ή και από τον υποψήφιο επίτροπο. Υπάρχει η διερμηνία σε 23 γλώσσες, επομένως όλοι μπορούν να χρησιμοποιήσουν την μετρική τους γλώσσα. Επενθυμίζω επίσης ότι όσα λέτε μεταφράζονται, ε, διερμηνεύονται και αυτό παρακαλείστε να μην μιλείτε πολύ γρήγορα. Επίσης μεταδίδεται από την ιστοσελίδα του Κοινοβουλίου ζωντανή η ε, συζήτηση, η ακρόαση και θα μπορέσετε να την δείτε, να την παρακολουθήσετε και αργότερα εφόσον μαγνητοσκοπείτε. Τα καθήκοντα που αναλαμβάνει ο υποψήφιο επίτροπος είναι πολύ σημαντικά. Δημοσιονομική σταθερότητα, δημοσιονομική ολοκλήρωση, αξιοπιστία των αγορών και αποτελεσματικότητα. Αυτά είναι και τα κέρια ζητήματα της σημερινής ακροάσεως. Επίσης βέβαια η ολοκλήρωση της Τραπεζικής Ένωσης, Ένωση Κεφαλαίου Αγορών για την διασφάλιση των επιχειρήσεων στην, ε, της, της πρόσβασης των επιχειρήσεων σε ε, χρηματοδότηση και αναμένουμε βέβαια μεγάλο ενδιαφέρον της απόψεις του υποψηφίου Επιτρόπου. Παρακαλώ κύριε υποψήφιε Επιτρόπου.